Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε ε, την συνεδρίασή μας με το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Γιάνν Κόχο, τη Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας και ασκούνται την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου ΓΚΑΕΡΚ, δηλαδή Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, που έλαβε χώρα χθε και σήμερα 23 και 24 Φεβρουαρίου. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Επιτροπή μας. Είμαστε πάλι γνώριμοι και περιμένουμε με περιέργεια και ανυπομονησία τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ασχολήθηκε και με τα Βαλκάνια. Ε, και εμείς ε, κατά σύμπτωση εξετάσαμε την ε, καταπληκτική έκθεση της Άννας Ιμπρισάτζιτς για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, τι γίνεται με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, θα διοριστεί νέος επιτετραμένος. Τι γίνεται με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Έχει πιθανότητες ένταξης. Τι γίνεται με το Κωσυφοπαίδιο και την ανάπτυξη της δύναμης Ulex. Τι γίνεται με την εταιρική σχέση με τη Σερβία, πώς ε, βαίνουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το Ερεινό Συμβούλιο. Φυσικά ένα από τα λάβαρα της Τσεχικής Προεδρίας είναι η ανατολική σχέση γειτονίας Ε, βέβαια αφημολογούνται διάφορα για το θέμα αυτό και πώς θα συνδυαστεί με τη συνέργεια για τον εύξηνο πόντο. Επίσης έχουμε το θέμα της ενέργειας και του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Έχετε το λόγο κύριε Προεδρεύοντα, θα ακολουθήσει γύρω σε ερωταπαντήσεων. Σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Καλωρίζει και κοινή αίθουσα. Θυμάμαι την περασμένη φορά ε, συνεδρίας παρουσίασα ε, τις θέσεις μου σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Αυτή είναι η τρίτη. Χαίρομαι για τις νέες αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας ενημερώσω εντάχει για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γκάρ, Κοινικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων και για τις αποφάσεις που έλαβε. Και φυσικά περιμένω τις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας για τη συζήτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σας αναφέρω εν συντομία δύο πολύ σημαντικά θέματα από την οριζόντια διάσταση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και την προετοιμασία για το Εωρινό Συμβούλιο του Μαρτίου. Τρία ήταν τα βασικά σημεία. Καταρχήν αναφερθήκαμε στην ε, διάταξη των εργασιών, περισσότερο στον τύπο παρά στην ουσία. Τα θέματα του Ευρωπαϊκού Ερνού Συμβουλίου θα είναι η οικονομική και δημοσιονομική χρηματοπιστωτική κατάσταση, θέμα κλιματικών αλλαγών, τρίτο εξωτερικές σχέσεις και τέταρτο συνθήκη της Λισαβόνας. Χθες επίσης ασχοληθήκαμε με το πολύ σημαντικό θέμα το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προγράμματα που καλύπτει και τη χρηματοδότησή του. Φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει ήδη για ορισμένα από τα συμπεράσματα. Εκτενής ήταν και η συζήτηση για τα επιμέρους σχέδια του σχέδιου αυτού και το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν έχει αριστικοποιηθεί όμως η απόφαση. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για τα περισσότερα από τα σχέδια, τα επιμέρους σχέδια του σχεδίου ανάκαμψης. Και επίση εκκρεμούν ορισμένε πτυχές της χρηματοδότησης του. Ευελπιστούμε πάντως ότι μέχρι το Μάρτιο θα είμαστε έτοιμοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να διεκπαιρεωθούν όλα αυτά τα θέματα. Έγινε μία σύντομη συζήτηση και τη ημερήσια διάταξη αυτού του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ασχοληθεί με τα ίδια θέματα που θα απασχολήσουν και το επίσημο Ερεινό Συμβούλιο προκειμένου να προλιαθεί κάπως το έδαφος και να βολιδοσκοπηθούν τα κράτη-μέλη για το ποια είναι τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να γίνουν και οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. και να δούμε προς τα πού θα στραφεί περισσότερο η συζήτηση του επίσημου Ειρηνού Συμβουλίου. Όλα αυτά θα απασχολήσουν το προηγούμενο άτυπο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ε, εγκρίναμε τα συμπεράσματα για τη Σρι Λάγκα. Ζητήσαμε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και του πυρός, προκειμένου να διοχετευθεί απρόσκοπτα η ανθρωπιστική βοήθεια και μετά τις εξέλιξεις περασμένης εβδομάδας καταδικάσαμε δρυμύτατα τις ε, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας ε, στο Κολόμπο το Φεβρουάριο που είχαν ε, πολλά θύματα και τραυματίες. Υιοθετήσαμε τα συμπεράσματα και για το Ιράκ μετά τις τελευταίες εκλογές και πάλι εκφράσαμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαδικασία εκδημοκρατισμού και σταθεροποίησης στο Ιράκ. Κατά τη συζήτηση για το Αφγανιστάν σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει κατεπηγόντως να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς το λαό και την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και θα έχουμε τη διαδικασία αναθεώρησης της συμβολής μας στο Αφγανιστάν που θα πρέπει να επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική. Το Αφγανιστάν θα αντιμετωπίσει πολύ σημαντικές προκλήσεις τον υπόλοιπο χρόνο με ένα μισή χρόνο. Ιδιαίτερα έχουμε τις επικείμενες εκλογές που θα σηματοδοτήσουν τις επόμενες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και την νομιμοποίηση της ε, επόμενη κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για τη χρηματοδότηση των εκλογών και θα αναπτύξει μια πολύ σημαντική πολυμελή αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον συντονιστικό ρόλο της ε, αντιπροσωπείας του ΟΗΕ στο, στο Αφγανιστάν και τον ρόλο παρατήρηση που θα διαδραματίσουν για τι εκλογέ. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την αποστολή Γιούπολ στα πλαίσια της νέας στρατηγικής. Επίσης θα πρέπει να επικουρήσουμε τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους του Αφγανιστάν. Η σωστή αστυνόμευση είναι χέγγιο της σταθερότητας στο Αφγανιστάν. Εκτός από τη Γιούπολ θα πρέπει να δούμε και άλλους τομείς στους οποίους θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τη θέμενη αξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ευρύτατες αρμοδιότητές της θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, θα επικεντρωθεί κυρίως στη διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Οι Υπουργοί συμφώνησαν και για τη σημασία ενός ευρύτερου περιφερειακού πλαισίου και μιας ε, πολύ ε, θετικής δέσμευσης και ανάμεξης των γειτονικών χωρών και άλλων παραγόντων του Αφγανιστάν η περιφερειακή προσέγγιση θα πρέπει να αντιμετωπίσει καλύτερα θέματα καταμερισμού του βάρους, ιδιαίτερα σε θέματα αντιτρομοκρατικού αγώνα και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών. Οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας με τις ΗΠΑ προκειμένου να βρεθεί κοινή προσέγγιση για τη σωστή εφαρμογή των λύσεων με στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και ισχυρότερου Αφγανιστάν. Γιατί, για το Μέση Ανατολικό συζητήσαμε την κατάσταση στο, στη Μέση Ανατολή προετοιμάζοντας την διεθνή διάσκεψη που θα γίνει στο Σαρμελσέ για την ανασυγκρότηση της Γάζας στις 2 Μαρτίου. Το βασικό μήνυμα της διάσκεψης αυτής θα είναι η συμπερίληψη της ε, προσπάθειας της Αιγύπτου στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες ανάγκη βοήθειας της Παλαιστινιακής και στήριξης Παλαιστινιακής Αρχής και ανάγκη ανοίγματο των, περασμάτων στη Γάζα προκειμένου να λάβει χώρα μια ουσιαστική ανασυγκρότηση και ανάκαμψη. Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Γειτονία που συζητήθηκε στη διάρκεια του γεύματος. Για πρώτη φορά τέθηκε το θέμα της Ανατολικής Γειτονίας στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Η συζήτηση έγινε προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο πολιτικός και στρατηγικός στόχος του προγράμματος. Υπήρξε γενική συνένεση ότι το θέμα της ανατολικής γειτονίας είναι βιώσιμο. Γι' αυτό και οι διαδικασίες σύνδεσης ε, βοηθούν στην ευάθυνση και στη δημιουργία κοινών ε, πλατφόρμων ε, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Οι Υπουργοί εξέτασαν το βαθμό συμβατότητας της ανατολικής γειτονίας με άλλες διαστάσεις όπως είναι τις συνέργειες για τον εύξηνο πόντο, θέματα, θέματα ελάφρυνσης των διατυπώσιο και τις θεωρίες και το καθεξής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο Συμβούλιο Κορυφής δήλωσε την επιθυμία του να δώσει μια, ένα σημαντικό περιεχόμενο στην Ανατολική γειτονία. Επίσης για το θέμα του διαρρισμού του νέου USR και την μεταβίβαση από το UHR στο USR συζητήθηκε επίσης. Έχουμε και το θέμα της υποβολής της υποψηφιότητας του Παυραβωνίου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρξε συνένεση για το θέμα αυτό. Θα το επεξεργαστεί περαιτέρω η Προεδρία τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης έγινε μια ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την ε, έναρξη εφαρμογή ε, της διάμεσης συμφωνίας με τη Σερβία. Υπό το φως όμως και των τελευταίων εξελίξεων στο Κωσυφοπαίδιο. Αυτά ήταν σε έδρες γραμμές ε, όσα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Να σας αφήσουμε λίγο χρόνο τώρα για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για αυτή την επισκόπηση. Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο αγορητή να πω ότι σημειώνουμε ότι η εταιρική σχέση αυτή με τι ανατολικέ χώρε είναι από του βασικού άξονε τη Προεδρία σα και συζητήθηκε η βάση του εγγράφου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που γνωρίζουμε και βάσει του εγγράφου τη Προεδρία και τη προόδου, εκθέσεω προόδου τη Προεδρία που δεν γνωρίζουμε, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα μπορούσε να ενημερωθεί. Θα μπορούσε να παραλάβει αυτά τα έγγραφα. Ερώτημα. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία Ιμπρεσεγκάτση. E, Ευχαριστώ πολύ. για την ε, παρουσίαση αυτή θα ήθελα να επενέσω και την Τσεχική Προεδρία και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε θέσει στις προτεραιότητά σας τα Βαλκάνια. Ίσως ε, καλύτερα θα ήταν να μιλήσω σου ειδικά, γιατί έκανα και την απόπειρα μου την πρώτη στα τσέχικα. Αναφέρεται λοιπόν ότι χτες ε, πώς διαμορφώθηκαν χθες οι προτεραιότητες. Ξέρω ότι η αίτηση του Μαυροβουνίου για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έγινε σχετική συζήτηση από, από ό,τι άκουσα και δεν ήταν θετική η τοποθέτηση. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα στοιχεία για το Μαυροβούνιο και το πώς ε, θεωρείτε εσείς ότι ως Προεδρία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Μαυροβούνιο. Πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθεί η κατάσταση με πιο θετικό τρόπο. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κ. Πλιμπετίτσο έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, κάτι να σκεφτούμε. Εδώ και ένα χρόνο το Κωσυφοπέδιο γινόταν ανεξάρτητο. Τώρα Κάποιες χώρες της Ενώσεως δεν αναγνωρίζουν αυτή την εξαρτησία. Ποια είναι η απόψη σας για αυτή την κατάσταση σαν Προεδρεύων του Συμβουλίου και τι απο, απολογισμό μπορεί να κάνετε για αυτό το έτος της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βιλόσοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά. Έχω δύο ερωτήσει κύριε Υπουργέ. Και, τα οι δύο αφορούν την ενέργεια. Η καταστροφή του Ιανουαρίου μπορεί να επαναληφθεί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επανάληψη αυτής της τραγωδίας και να έχουμε ένα κατάλληλο σχέδιο αντίδρασης. Η Ουγγαρία βοήθησε τελικά τη Σερβία, έδειξε μια ουσιαστική αλληλεγγύη και βοήθησε αποτελεσματικά υπήρξαν δυνατότητες, αλλά δεν βοήθησαν άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία, την Σερβία για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τσεχική Προεδρία είναι έτοιμες ε, να μας διαβεβαιώσουν ότι σε περίπτωση τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε πιο αποτελεσματικά. Και έχω και μία δεύτερη ερώτηση για τα ενεργειακά θέματα οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα, τι σκοπεύουν να κάνουν προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία που όπως μας λέει ο τύπος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά ε, την πώληση ενό από τα τελευταία σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του αγωγού φυσικού αερίου. Τέτοια ε, δυνατότητα εξετάζει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Τόσο δεινή είναι η χρηματοπιστωτική της και οικονομική της κατάσταση. Πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει κάπως στην ε, Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χόρατσεκ. Ehm, eh, Χαιρετίζω ξανά την τσεχική ε, προεδρία, μιλάω γερμανικά. Ε, eh- Χτες με την αντιπροσωπή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κροατίας βρέθηκα στο Ζάγκρεπ, στον Πρωθυπουργό Σάνοντα και στον Πρόεδρο Μέση, που επισκεφτήκαμε. Διαπιστώσαμε το πρόβλημα αυτό μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, το πρόβλημα αναφορικά με τα σύνορα, είναι πιο σοβαρό και με μεγαλύτερε συνέπειε από ό,τι φανταζόμαστε. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, τι σκοπεύει να κάνει η Τσεχική Προεδρία προ αυτήν την κατεύθυνση και τι κάνει ήδη. Και κατά δεύτερον, εν ώψη της επόμενης συνόδου με τη Ρωσία. Το Μάρτιο θα λάβει χώρα. Και θυμάμαι ότι εδώ και χρόνια θίγεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα για τους φίλους μας του Memorial, για τη νέα αγωγή κατά του Χοντογκόσκη και του Πλάτων και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η τσεχική προεδρία δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Thank Σας ευχαριστώ. Αυτός είναι ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Ο λόγος στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζω στα τσεχικά. Ναι, και είναι πολύ δημοφιλή γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω φάνηκε την περασμένη εβδομάδα. Στον αφορά το έτοιμά σα για το έγγραφο, για τα έγγραφα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα non-paper της ε, Προεδρίας. Οπότε θα μπορούσαμε να σας το δώσουμε. Και αυτό αναφέραμε και μπορούμε να σας το δώσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Όσον αφορά την έκθεση πρόοδου, είναι εμπιστευτικό, εμπιστευτικό έγγραφο αυτό, αλλά προφανώς αν αλλάξει το καθεστώς του και δεν είναι πια εμπιστευτικό θα μπορέσουμε να σας δώσουμε και αυτό το έγγραφο, την έκθεση στην Επιτροπή. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε από την Επιτροπή σας. Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, όπως ανέφερα προηγουμένως, ήταν μια συζήτηση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του γεύματος, απουσίαζα δυστυχώς, αλλά από ό,τι γνωρίζω, από αυτά που διάβασα, από το υλικό που ήταν στη διαθεσή μου διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει συνένεση. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια διαδικασία που θα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να παρουσιάσει μια γνωμοδότηση εντός 12, 14, 16 μηνών την άποψή της, την γνωμοδότησή της. Για την ώρα το Μαυροβούνιο αυτό καθεαυτό δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα θεωρηθεί η όλη κατάσταση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα κάποιες χώρες δεν θεωρούν το ζήτημα απλώς ένα τεχνικό ζήτημα που είναι η προσέγγιση που ακολουθεί η Προεδρία και οι περισσότερες χώρες. Αλλά θεωρούν ότι εντάσσεται αυτό το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ε, υπάρχει συνένεση αφορά τη διεύρυνση και προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνένεση για συγκεκριμένες χώρες και εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες, το έχουμε πάντα υπόψη μας το ζήτημα και θα το επανεξετάσουμε, θα το ξανασυζητήσουμε με τους διάφορους εταίρους και στο Συμβούλιο του Μαρτίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα το συζητήσουμε. Τι κάνει το Συμβούλιο όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν επίσημα το κοσυφοπέδιο Και επειδή αυτή είναι εθνική απόφαση, το Συμβούλιο και η Προεδρία δεν μπορούν να πιέσουν καμία χώρα. Είναι στην διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας αυτή η απόφαση. Αυτό που είναι κρίσιμο και όπου υπάρχει συμφωνία είναι το EULAX και οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του και οι ευρωπαϊκές προπτικές του Κωσυφοπεδίου και άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη επέτειος, στην πρώτη επέτειο, βλέπουμε ότι 57 χώρες έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο και αυτή είναι μια πολιτική πραγματικότητα. Και για μας και το Συμβούλιο αυτό που είναι σημαντικό όσον αφορά τις προοπτικές που ανοίγονται για τις χώρες αυτές. Υπάρχει συμφωνία δηλαδή για διεύρυνση προς τις χώρες Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα όσον αφορά την ενέργεια πρέπει να σας πω σχετικά με το θέμα αυτό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αποκατάστασης και τα διάφορα προγράμματα που έχουν υποβληθεί ως προτάσεις έχουν υποβληθεί σε αναθερημένη μορφή για δεύτερη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών αυτής κατά τη διάρκεια της κρίσης του φυσικού αερίου που διαπιστώσαμε πρόσφατα. Και σχετίζεται αυτό και με την διασύνδεση μεταξύ χωρών όπως είναι η Βουλγαρία, Ουγγαρία κλπ. Όμως δεν έχει επέθει συμφωνία στο Συμβούλιο όσον αφορά αυτά τα προγράμματα. Χρειάζεται μια γεωγραφική ισορροπία και χρειάζεται μια συμφωνία όσον αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος, αυτό είναι σίγουρο. Θέλουμε να υπάρχει ασφαλής εφοδιασμός ενεργειακός και όχι μόνο όσον αφορά το φυσικό αέριο αλλά και όσον αφορά άλλες μορφές ενέργειας. Η κατάσταση, το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί. Είναι οι κασίες αυτό ε, δεν αλλάξαν πολλά βέβαια από τον Ιανουάριο και αν ξανασυμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο όπως με το φυσικό αέριο θα ήταν παρόμοιο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει σε ένα φόρουμ που θα προσπαθήσει να προσελκύσει επενδυτές, οι οποίοι επενδυτές ίσως να χρηματοδοτήσουν αυτά τα διάφορα ε, συστήματα και δίκτυα διελεύσεως ε, της ενέργειας διελεύσεως και μέσω της Ουκρανίας, ούτως ώστε να διατηρηθεί ο ασφαλής εφοδιασμός και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ουκρανίας. Προφανώς τα ουκρανικά οικονομικά προβλήματα και της Ανατολικής Ευρώπης, αυτά τα οικονομικά προβλήματα ε, δυσκολεύουν την κατάσταση και βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν προβλήματα, τα βλέπουμε στον τύπο. Βέβαια οι αναφορές στον τύπο είναι κάπως υπερβολικές. Κατά την άποψη της Προεδρίας η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες και αυτό πρέπει να συζητηθεί 1η Μαρτίου και μετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μετά την 1η Μαρτίου. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Τσεχικής Προεδρίας, όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ Σλοβενίας και ε, Κροατίας, τη διένεξη που υπάρχει, πρέπει να σας πω ότι σαν Προεδρία προσπαθούμε να είμαστε πολύ διακριτικοί, προσπαθούμε να διευκολύνουμε την εξομάλυνση του ζητήματος αυτού που είναι βασικά διμερούς χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε και αυτή να συμμετάσχει στις προσπάθειες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιο χώρο ε, συζήτησης και κατανόησης και επίλυσης του προβλήματος το ταχύτερο δυνατόν και να βρεθεί και μια λύση ικανοποιητική και για τις δύο χώρες ούτως ώστε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία να μπορέσουν να συνεχιστούν ε, με κανονική ταχύτητα δεν είναι αποκλειστική η δραστηριότητα αυτή της τσεχικής προεδρίας, είναι μια προσπάθεια που καταβάλλεται και μέσω διαπραγματεύσεων και συμβολής και άλλων. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συζητήσεις της Σύνοδο Κορυφής με τη Ρωσία, η τσεχική προεδρία μπορεί να σας υποσχεθεί ότι θα είναι στο πρόγραμμα αυτό το θέμα και θα συζητηθεί. Σας ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Πρώτη ερώτηση δική μου. Συναντήσα, ενημερώσατε, συναντήσατε και τον κύριο Χαβιέ Σολάν, ενημερωθήκατε τις επισκέψεις του στο Μίνσκ, στη Λευκορωσία. Τι έγινε. Ο κύριος Κυρίλοφ θέλει επίσης να υποβάλει μια ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό και από τους προλαλήσαντες. Με ευρώντητος από το ότι δεν συζητήθηκε σχεδόν τίποτα για την γενική οικονομική κατάσταση. Γίνεται λόγος για ανάκαμψη και αναφερθήκατε στο σχέδιο ανάκαμψη, αλλά βλέπετε τι γίνεται γύρω μας και πόσο δεινή είναι η κατάσταση οικονομική. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους σχέδια που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, Εντάξει, αυτά είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και απτά. Εμένα με ενισχύει περισσότερο η κατάσταση που επικρατεί γενικά και το, ο κίνδυνος γενικής αποσταθεροποίησης, οικονομικής που ολοχεύει σε ορισμένες χώρες. Εντάξει, σίγουρα δεν απειλούνται όλε οι χώρε από μια τέτοια αποσταθεροποίηση οικονομική, αλλά το τραπεζικό σύστημα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ανήκει σε αλλοδαπέ τράπεζε. και η πολιτική του πίστοσης, χορήγηση πίστοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άνηση δανεισμού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά αποτελέσματα γιατί υπάρχει αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση, κάτι που θα επιδεινώσει το γενικό οικονομικό περιβάλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε κάποια κρούσματα προστατευτισμού και δημόσιες δηλώσεις που έγιναν σε κάποιες χώρες υπέρ του προστατευτισμού. Με ενδιαφέρει λοιπόν ε, αν συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Καλές οι τυπικές, οι επίσημες, οι άτυπες συνεδριάσεις. Το θέμα αυτό όμως συζητήθηκε, το θέμα της οικονομικής κρίσης συζητήθηκε στο Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, γιατί πραγματικά αυτό το θέμα απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος Μιγιαν Σα ευχαριστώ. Εγώ θα ασχοληθώ κυρίως με δύο θέματα, κύριε Υπουργέ. Στο πρώτο αναφερθήκατε κι εσείς ακροθυγός. Σε ό,τι αφορά τη συνδιάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ποια είναι η... ποιο είναι το ποσό που εξετάζει το Συμβούλιο για την ευρωπαϊκή αρρωγή. Έχετε κάποια ιδέα για το σε τι ποσό θα ανέλθει αυτή η ευρωπαϊκή συνδρομή για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ήδη. Μπορείτε να μας τα δώσετε για να τα συγκρίνουμε με τις συνεισφορές των υπόλοιπων παγκόσμιων εταίρων. Για να δούμε ποια θα είναι η σχέση της δικής μας συνδρομής με τη συνδρομή των υπολείπων δωρητών. Να κάνουμε μια συγκριτική εξέταση. Δεν ξέρω αν το συζήτησε χθε σήμερα το Συμβούλιο, αλλά εμεί σήμερα εξετάσαμε και εγκρίναμε μάλιστα μία έκθεση για τις διατλαντικέ σχέσεις. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδε αν δεν κάνω λάθο, η εκπρόσωπο τη Τσεχική Προεδρίας συνάντησε την ε, Αμερικανίδα Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Χίλαρη Κλίντον. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα από την ε, συνάντηση αυτή. Τον Απρίλιο θα υποδεχθούμε στην Ευρώπη τον πρόεδρο Ομπάμα για την 60η επέτειο του ΝΑΤΟ. Τι προοπτικές υπάρχουν, θα, θα γίνει κάποιο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σαν αυτό που έγινε στις 25 Φεβρουαρίου του 2005 με τον Μπούς. Θα έρθει ο κύριος Ομπάμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι προοπτικές υπάρχουν για την επίσκεψη του Πρόεδρου Ομπάμα στην Ευρώπη. Τι σχέδια έχει το Συμβούλιο, τι οράματα για, την, για επαφές με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ναζαρέ. ναι, έχω εντυπωσιαστεί. Δύο ρωτήσεις. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη μείωση της χρηματοδότηση για τον Αμπούκο από 250 εκατομμύρια σε 200 εκατομμύρια, το οποίο συνέβη λίγες εβδομάδε μετά την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να επιταχύνει το project. Αναρωτιόμουν μήπω αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ω έλλειψη συνοχή σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Και επίση, αν δεν δεν αποστέλνει αρνητικά μηνύματα για το συγκεκριμένο project αυτή η μείωση τη χρηματοδότησης. Επίση να ρωτήσω κατά πόσο μια αρχική δέσμευση αναφορικά με το project ε, του Ναμπούκο. Εξακολουθεί να είναι η ίδια σε αυτό το τροποποιημένο ε, πλαίσιο που ουσιαστικά έχει γίνει περικοπή 50 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλήσατε για το φόρουμ των επενδυτών που θα δαπανίσουν χρήματα για ενεργειακά προγράμματα. Αν μήπως δίνουμε αρνητικά μηνύματα προς αυτούς τους ξένους επενδυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά αυτά προγράμματα τα οποία παρουσιάσατε, θα μπορούσατε να κάνετε μία αξιολόγηση για το τι ποσοστό των προγραμμάτων αυτών έχει για τι ποσοστό των προγραμμάτων αυτών έχει γίνει η μελέτη εφικτότητας και κατά πόσον είναι σε θέση να εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά αν υπάρχουν διαφορές ε, αναχώρα και πώς διαχειρίζεστε αυτές τις διαφορές ενδεχομένως. Σας ευχαριστούμε κύριε Ναζαρέ. Αυτό ήταν ο δεύτερος λόγο. Γύρω σε ερωτήσεων, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να επανέλθω στο δικό σας το ερώτημα που θέσατε. η Λευκορωσία ως θέμα δεν τέθηκε στο Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Τέθηκε στις ε, γενικότερες, ε, στο πλαίσιο των γενικότερων διαπραγματεύσεων και όπως ξέρετε συνεχίζονται οι συζητήσεις για το κατά πόσο θα συμμετείχε και με τη ιδιότητα Λευκορωσία στην αρχική αυτή σύνοδο. Σημείο αφετηρίας μας και αυτό το είπα και στην προηγούμενη συνάντησή μας, μετά την συνάντηση της Τρόικα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας, το Συμβούλιο θα ξαναξετάσει την αναστολή των κυρώσεων στην συνάντηση του Απριλίου. Και εν τω μεταξύ θα εξετάζουμε τον κατάλογο που μας έδωσε ο κ. Μάρτινοφ για να δούμε που έχει επιτευχθεί προοδός. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε με τη Λευκορωσία μας προκαλούν μεγάλη σύγχυση. Ωστόσο, και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα συμπεράσματα. Ο Χαβιέ, τα συμπεράσματα που παρουσίασε ο Χαβιέ Σολάνα, η ηγεσία της Λευκορωσίας αντιλαμβάνεται πως έχει η κατάσταση και καταλαβαίνει ποιο είναι το διακύβευμα. θα ήθελαν και αυτοί να συμμετέχουν στην ε, ευρωπαϊκή γειτονία και κάτι το οποίο ακούσαμε για την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση και κάτι αυτό το ακούσαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που θα προκαλούσε μεγάλη σύγχυση θα ήταν αν η Ρωσία αναγνώριζε την Εμφχαζία και την Νοτιοασυντία. Γι' αυτό ο Χαβιέ Σολάνα μας μετέφερε το μήνυμα ότι η ηγεσία κατανοεί ότι κάτι θα πρέπει να πράξει και ότι θα ήθελαν όντως διακαώς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση της συζήτησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γενικότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση αυτή, ίσως να επικρατεί και κάποια σύγχυση γιατί γίνεται τεράστιος αριθμός διαδικασιών, συναντήσεων, συνόδων. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ε, αυτές για την προετοιμασία του G20 ή τη Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τσεχική Προεδρία θα ήθελε να τα δει όλα αυτά συνολικά και να τα συζητήσει από κοινού. Το Συμβούλιο αυτό Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων δεν προσπάθησε να εξεύρει λύσεις, γιατί αυτό εξαρτάται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και από τους Πρωθυπουργούς. Εμείς προσπαθήσαμε να θέσουμε την ατζέντα και όπως σας είπα, αυτή η ατζέντα έλαβε την υποστήριξη όλων. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση στο Μαϊλίν, ένα από τα σημαντικά μηνύματα ήταν η ανάγκη καταπολέμησης του προστατευτισμού. Αυτό μας ε, το λένε και πρέσβεις και εκπρόσωποι διάφορων διεθνών οργανώσεων ανά τον κόσμο. Έχω συνδεθεί με πολλούς εξ αυτών τις τελευταίες εβδομάδες. Αποτελεί πραγματικά ένα δρόμο χωρίς γυρισμό. Και έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και τη ρύθμιση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγοράς και σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των προϊόντων τους. Αυτό θα συζητηθεί κατά την προετοιμασία της ενεπίσημης συνόδου. Στην 1η Την 1η Μαρτίου η Τσεχική Προεδρία θα επικεντρωθεί στα θέματα αυτά και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει σαφή συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν και τις κατευθυντήριες γραμμές για όσους θα συμμετάσχουν στη συνάντηση του G20. Και είναι σαφές ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν την αίσθηση ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με μία κοινή φωνή. Γιατί πρόκειται για μία πολυτέλεια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να δράσουμε. Δηλαδή ε, ο καθένας για τον εαυτό του. Τώρα σε ό,τι αφορά την Γάζα, δυστυχώς δεν έχω τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Αναφορικά με τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, γιατί σε ό,τι αφορά... Δεν, δεν συζητήσαμε ακριβή ποσά. Θα συζητηθούν συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με την παροχή βοήθειας, τον πρόεδρο Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, την υποστήριξη προς την Αίγυπτο και τις ε, διαδικασίες ε, τις σχετικές ε, με τις διαπραγματεύσεις. Ε, Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Ιστορικών Σχέσεων δεν ε, συζήτησε τις διατηρητικές σχέσεις και την, την πρόθεση πρόσκλησης της κυρίας Κλίντον. Ωστόσο, γίνονται ανεπίσημες συζητήσεις και όπως ξέρετε η Τσεχική Προεδρία θα χαιρόταν να διοργανώσει συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ομπάμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 27 κατά την επισκέψή του στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια τέτοια συνάντηση. Όταν λοιπόν ε, λάβουμε τα ανάλογα μηνύματα θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε. Αλλά βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή η πιθανότητα να γίνει μια τέτοια συνάντηση αυξάνεται. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς την κατεύθυνση αυτή ωστόσο. Αναφορικά με την ε, Μείωση της χρηματοδότησης για τον αγωγό του Ναμπούκο από 250 εκατομμύρια σε 200 εκατομμύρια. Όπως σας είπα, ο κατάλογος των προγραμμάτων και ο τρόπος χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών είναι κάτι το οποίο δεν έχει λάβει την οριστική του διαμόρφωση. Ξέρετε ότι το αρχικό ποσό, τα 3,5 δισεκατομμύρια για τα project αυτά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project και τα project διαλειτουργικότητας, έχει αυξηθεί το αρχικό ποσό από 3,5 σε 3,75 δισεκατομμύρια. Και κατά τις ε, συζητήσεις μας για τα project αυτά, ε, ακούστηκαν διάφορα σχόλια. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ενός πιο ισορροπημένου, ενός πιο σταθεσμισμένου καταλόγου προγραμμάτων η μείωση αυτή αποτελεί κάτι που δεν μπορεί να πω ότι αποτυπώνει την πολιτική διάθεση. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όπως σας είπα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε ό,τι αφορά τώρα τις μελέτες εφικτότητας. Πρόκειται για πολιετή προγράμματα κάποια εκ των οποίων ε, ενδεχομένως να ολοκληρωθούν φέτος, κάποια άλλα ίσως και στα επόμενα έτη. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα, ε, για όλα υπάρχει μελέτη εφικτότητας. Ωστόσο τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί επί πολλά έτη και δεν είναι πραγματικά προγράμματα τα οποία προέκυψαν εκ των Ουγκάνευ είναι πολύ σημαντικά και τα χρειαζόμαστε για την πραγματοποίηση της ε, ενιαίας αγοράς στον τομέα της ενέργειας και για να βελτιώσουμε και την ενεργειακή μας ασφάλεια και την διαλειτουργικότητά μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λίγο, Πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διεξοδική ανάλυση. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι στο Γκάρκ, Ευχαριστώ που ήθελα να μας ενημερώσετε. Πέρασε συνεδριά σας. Ευχαριστώ.